Δεν βλέπω να υπάρχουν, αλλά τα πρακτικά εγκρίνονται. Θέλω να ενημερώσω το Σώμα ότι μετά την ε, διακοπή της συνεδρίασης του Κοινοβουλίου στις 18 Απριλίου, ο Πρόεδρος και ο Πρόεδρος του, ο του Συμβουλίου υπέγραψαν 48 νομικά κείμενα που εγκρίθηκαν στα πλαίσια της ε, συνήθους νομοθετικής διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 78 του κανονισμού του Κοινοβουλίου. Οι τίτλοι των νομικών αυτών ε, πράξεων θα δημοσιευθούν στα πρακτικά της σημερινής συνεδριάσεως. Με βάση την ημερήσια διάταξη προχωρούμε στην εκλογή των αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να σας ενημερώσω ότι έλαβα τις ακόλουθες υποψήφιες Μπάρλι, Μπέρ, Πιτζότο, Καστάλντο, Τσαράζοβα, Ντόμπρεβ, Χάουταλα, Ουταζάρη, Γιάδοκα, Κάρας, κολάγια Κόπατς, Κρασνοντεύσκη, Μακκίνες, Παπαδημούλης, Σίλβα Περέιρα, Βίλαντ. Οι υποψήφοι επιβεβαίωσαν ότι δέχονται τις προτάσεις υποψηφιότητά τους, οπότε ξεκινούμε την ψηφοφορία. Η ψηφοφορία σε, στην πρώτη διαδικασία εκλογής. Να σας πω και κάποιες τυπικές διαδικασίες. Πρώτον, οι ψηφολέκτες είναι οι ίδιοι με αυτούς που ανέλαβαν τη διαδικασία για την εκλογή του Πρόεδρου. Παρακαλώ να έρθετε στις κάλπες. Είναι όλοι παρόντες. Λείπει κάποιος. Έρχεται η συνάδελφος Φίλιπς. Κάποιος άλλος. Είναι όλοι παρόντες. Allora, Δεν υπάρχει ενημέρωση απουσιών. Προχωρούμε λοιπόν οι ψηφολέκτες θα ψηφίσουν τελευταίοι. Επειδή ο αριθμό των υποψηφίων είναι υψηλότερο του αριθμού των θέσεων, θα πρέπει να προχωρήσουμε σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού μας σε μια ψηφοφορία με μυστική ψηφοφορία. Σας υπενθυμίζω τη σχετική διάταξη. Προχωρούμε διαδοχικά στην εκδογή με μία ψηφοφορία των αντιπροέδρων. Εκλέγονται στο πρώτο στον πρώτο γύρο έως 14 βουλευτές με την σειρά των ψήφων που έλαβαν. Οι υποψήφοι που έλαβαν την απόλυτη ε, πλειοψηφία των ψήφων που έχουν εκφραστεί. Αν ο αριθμός των εκλεγέντων είναι μικρότερος του αριθμού των θέσεων, προχωρούμε σε δεύτερο γύρο με την ίδια διαδικασία για την ανάθεση των υπόλοιπων θέσεων αντιπρέδρων. Εάν χρειαστεί τρίτη ψηφοφορία η εκλογή γίνεται με σχετική πλειοψηφία για τις υπόλοιπες θέσεις. Σε, περίπτωση, σε περίπτωση ισοψηφίας κηρύσσεται εκλεγής ο υποψήφιος, ο, ο αρχαιότερος υποψήφιος. Σας διανέμονται... Γκέτα, ο συνάδελφος Γκέτα πρέπει να πάει στην κάλπη LM. Γετά. Πρέγω, Εσέντσι δε ρεγολαμέντο. Ε, επί του κανονισμού ζητάτε το λόγο. Ναι, Πρόεδρε, 61% των Ευρωβουλευτών είναι καινούργοι. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί οι υποψήφοι αντιπρόεδροι. Δεν μπορεί να υπάρξει μια δήλωση σύντομη από τον καθένα εξ αυτών γιατί είναι υποψήφιοι. Γνωρίζω κάποιους από τη δική μου ομάδα, αλλά από τι άλλε ομάδε δεν του γνωρίζω. Η παρατήρησή σα, μου επιτρέπει να θυμίσω ότι η διάσκεψη των πρόεδρων αποφάσισε ότι αυτό θα επιτρέπεται μόνο στους υποψηφίους για τη θέση του Προέδρου και όχι του Αντιπροέδρου. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο δεν κατέστη δυνατόν να, μπουν, να μπει αυτή η διαδικασία στην μερίσια διάταξη. Παρακαλώ τους κλητήρε να ολοκληρώσουν την ε, διανομή των ψηφοδελτίων και των φακέλων. Σας ε, υπενθυμίζω ότι οι θέσεις είναι 14, άρα ο κάθε βουλευτής μπορεί να δώσει έως 14 επιλογές. Σας θυμίζω ότι πρέπει να ψηφίσετε τουλάχιστον 8 υποψηφίους. Αλλιώς το ψηφοδέλτιό σας θα θεωρηθεί άκυρο. Βεβαίως δεν μπορείτε να υπερβείτε τον αριθμό των 14 προτιμήσεών σας. Γιατί και σε αυτή την περίπτωση το ψηφοδέλτιο θα θεωρηθεί άκυρο. Άρχεται η ψηφοφορία. Και περιμένουμε πλέον την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας. Allora, la η ψηφοφορία και παρακαλώ τους ψηφολέκτες να προχωρήσουν στην καταμέτρηση. Διακόπτεται η συνεδρίαση. Θα ενημερωθείτε όσοι ήθιστε από το καμπανάκι για το πότε θα ξεκινήσουμε. Και θα το δείτε και στις οθόνες. Διακοπή συνεδριάσεως.